τα πρακτικά. Διακόπτουμε λοιπόν την συνεδρίαση και ευχαριστώ όλους για την παρουσία τους εδώ. Τον Επίτροπο που ήρθε, τους διερμηνείς. Καληνύχτα. Αν καλό φαγητό, αλλά υπάρχει και μια πολωνική παροιμία. Πρωινό μόνος, μεσημέρι με τους φίλους, βραδινό τους εχθρούς.